Έχω λάβει σε πρώτη ανάγνωση δύο θέσεις του Συμβουλίου, τον κανονισμό για τα ιατρικά προϊόντα, καθώς επίσης τον κανονισμό για τα διαγνωστικά in vitro. Θα δημοσιευθούν στα συνοπτικά πρακτικά οι τίτλοι και το Κοινοβούλιο διαθέτει τρεις μήνες για να ε, αποφανθεί. Η προθεσμία αρχίζει αύριο